Eh, Από την ε, ομάδα του Λαϊκού Κόμματος έχουμε πάρει τις εξής τροποποιήσεις στους ε, διορισμούς ε, μελών σε επιτροπές. Επιτροπή Αναφορών. Η κυρία Ματσόνη αντικαθιστά την κυρία Γκαρντίνη. Στην Επιτροπή Οικονομικών Μεταφορών. Η κυρία Ντεβεϊράκ αντικαθιστά τον κύριο Ρικέ. Από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών έχουμε λάβει τους εξής διορισμούς για τις κοινωνικές επιτροπές. Επιτροπή Αναφορών, η κύριοι Καμίνσκι και Κίρκχοπ. Επιτροπή Περιβάλλοντος, η κυρία Τσεσκόβα. Επιτροπή α, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κύριος Χέλμερ. Επιτροπή Ελευθεριών, ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ. Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναίκας, ο κύριος Κίρκχοπ. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κύριος Ντέβα. Και η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, ο κύριος Λεγκούτκο. Περνάμε στις ε, προτάσεις ε, ορισμού μελών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεν έχει υποβληθεί καμία τροποποίηση, καμία αλλαγή. Συνεπώς, ε, θεωρώ εγκεκριμένες τις προτάσεις της διάσκεψης των Πρόεδρων. Señora Harms,